Madame le Président. Bonjour à tous. Καλημέρα. Καλωσορίσατε στην Ολομέλεια. Προβλέπουμε σήμερα την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την κατάργηση του γυναικείου σεξουαλικού ακροτηριασμού και θα δώσω πρώτα πρώτα το λόγο στην κυρία Ζουμπέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε.